Σας ευχαριστώ. Αγαπητοί συναδελφοί, σε δύο εβδομάδες υπάρχουν βουλευτικές εκλογές στη Λευκορωσία. Εδώ και καιρό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρακολουθεί με προσοχή και ανησυχία τις εξελίξεις στην ε, χώρα αυτή και με ενισχύα βλέπουμε να συνεχίζονται οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του κράτους δικαίου και των δημοκρατικών αξιών. Κάποια γεγονότα είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά μεταξύ των οποίων η απαγόρευση ταξιδιών στο εξωτερικό για κάποιους πολιτικούς της αντιπολίτευσης και ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Με βάση ε, νόμους ε, που διευρύνουν τις δυνάμεις της, ε, και τις εξουσίες της ΚΑΓΕΜΠΕ. Και βέβαια είχαμε και την ε, απέλαση του Σουηδού πρέσβη. Ζητάμε λοιπόν όλοι από τον δικτάτορα μεταρρυθμίσεις και πολιτική αλλαγή. Και θα ήθελα εδώ πέρα να πω ξεκάθαρα ως μήνυμα προς αυτή τη χώρα. Πρώτο βήμα πρέπει να είναι η άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων συνεχιζόμενη κράτηση των Άλες Μπιαλίτσκι, Μιχάλη Στάτκεβιτς, Πάβελ Σεβιάρινετς, Σιάρη Καβαλένκα και Δημήτρη Ντασκέβιτς και άλλων πολλών πολιτικών κρατουμένων δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί. Σας το λέω εδώ πέρα γιατί πρέπει να γνωρίζουν αυτοί οι άνθρωποι πως δεν τους ξεχάσαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχει ένα θεσμικό όργανο που παλεύει για αυτούς και είμαστε εμείς. Ζητάμε λοιπόν από την κυβέρνηση να διασφαλίσει πώς τις βουλευτικές εκλογές θα τηρηθούν όλες οι διεθνείς προδιαγραφές και θα έχουν μια ευκαιρία όλοι οι υποψήφοι και θα μπορέσουν επίσης και οι παρατηρητές του ΑΣΕ να ασκήσουν το έργο τους. Επιπλέον, να σας ενημερώσω πως στις 30 Αυγούστου απέστειλα ε, μια επιστολή στον πρόεδρο της Δημοκρατίας της Γάμπιας μετά την εκτέλεση εννέα ατόμων. 25 χρόνια υπήρχε μορατόριο ε, για την θανατική ποινή στην ε, Γκάμπια. Γιατί βεβαίως η συνεργασία μας με τη χώρα αυτή βασίζεται στην υποχρέωση σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων και στην επιστολή μου ζήτησα από την κυβέρνηση αυτή να μην προχωρήσει σε περαιτέρω εκτελέσεις ανθρώπων και να εφαρμόσει το μορατόριο της θανατικής ποινής γιατί σε ένα κράτος το οποίο το ίδιο το κράτος σκοτώνει και αποφασίζει για τη ζωή και το θάνατο, δεν επικρατεί δικαιοσύνη αλλά εκδίκηση. Αυτή είναι η βαθύτατη πεποίθησή μας και γι' αυτό βεβαίως θα συνεχίσουμε να παλεύουμε. Κυρίε και κύριοι, εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ήδη ε, το έκανα γραπτός και θα ήθελα να το πω και εδώ πέρα, να συγχαρώ τον ε, συνάδελφό μας και πρώην αντιπρόεδρο τον Σταύρο Λαμπρινίδη για τον ορισμό του ως ειδικού απεσταλμένου για τα ανθρώπινα δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωρίζετε όλοι τον κύριο Λαμπρινίδη όχι μόνο ως ε, αποτελεσματικό στη διεξαγωγή των ψηφοφοριών εδώ μέσα αλλά με την εμπειρία του με την ε, εκπαίδευσή τους νομικός, με τις γνώσεις τους και με την ε, προσωπικότητά του νομίζω πως είναι ο κατάλληλος για αυτή την δουλειά και χαίρομαι που και εσείς συμφωνήσατε μαζί μου και από Λεμάνια της ε, στήριξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο κύριος Λαμπρινίδης. Οι αρμόδιες κυπριακές αρχές μου είπαν πως ε, ο κύριος Σοφοκλής καταλαμβάνει την θέση του κυρίου Κυριάκου Μαυρονικόλα από